Good morning Καλημέρα σας. Ας αρχίσουμε και πάλι λοιπόν. Ανακοινώσει του Προέδρου. Διορισμοί εισηγητών ε, συντακτών γνωμοδότης από τη χθεσινοβραδινή η απογευματινή συνεδρίαση των συντονιστών. Starting with the nomination of rapport. Διορισμός εισηγητών για τις βασικές νομοθετικές εκθέσεις πρόταση οδηγίας για υποδομή εναλλακτικών καυσίμων από το ΕΛΚ. Κάποιος θα αναλάβει την έκθεση. Πρόταση κανονισμού για την αντικατάσταση του κανονισμού 1192 σχετικά με τους σιδηροδρόμους στην ΚΟΕ. Πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Σιδηροδρόμων ε, ε, και αντικατάσταση του 881 συντηρητική πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό 13-17 για τη διάνοιξη των αγορών για εγχώριες σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών το ΕΛΚ πρόταση οδηγία που τροποποιεί την 34 του 2012 που ε, δημιουργεί ένα ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο και φορά τη διάνοιξη των αγορών και πάλι ε, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σε χώριες και τη διαχείριση των υποδομών των μεταφορών σιδηροδρομικών ε, το παίρνουν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πρόταση οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα των σιδηροδρομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή φιλελεύθερη πρόταση οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στους πρασίνους μη νομοθετικές εκθέσεις τώρα. Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υπογράφουν, κυρώνουν ή να ε, προσχωρούν στη Συμφωνία της Cape Town το 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλου που σχετίζεται με τη διεθνή ε, σύμβαση του Τορεμολίνος για τα ληφτικά σκάφη Άλντε. Η φιλελεύθερη για το έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την οδηγία 1999-62 ε, για βαρέα οχήματα αποφάσισαν οι συντονιστές να μην αναλάβουμε δράση καθόλου. Είναι απλώς ένα έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις νομοδοτήσεις τώρα. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για το πρόγραμμα δράσης 2020 για τις επιχειρήσεις. Καμία δράση δεν θα έχουμε εμείς το έγγραφο εργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα που θα ανταλλάζουμε πληροφορίε για το περιβάλλον Outlook, καμία δράση, για το CARS 2020 πρόγραμμα δράσης για μια αυτοκίνητο βιομηχανία βιώσιμη ε, και ανταγωνιστική γνωμοδότηση που θα πάρουν οι συντηρητικοί ECR, προτεραιότητες για το προπολογισμό ε, του 2014 τμήμα 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότηση πράσινη γιατί έχουμε ένα κανονικό πάγιο σύστημα εναλλαγής των ε, εισηγητών για τον προπολογισμό. Συνιστούν επίση οι συντονιστέ να μην αναλυφθεί η δράση ω προ την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Καθαρή Ενέργεια για την τέταρτη δέσμη μέτρων για τα σιδηροδρομικά. Και τις σχετικές ανακοινώσεις για το υπόλοιπο τέταρτο πακέτο. Μην ακρόαση για το καμποτάζ στο σιδηρόδρομο αποφασίστηκε να διοργανώσουμε μήνυα ακρόαση με συμμετοχή επιλέκτων ενεχομένων πριν ε, υποβληθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα συνδυαστεί με τις παρουσιάσεις των δύο μελετών που έχουμε αναθέσει για την ανάπτυξη και εφαρμογή του καμποτάζ του σιδηροδρόμου στην Ένωση και τις ε, εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες ε, των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο. Επιτροπολογία. Σημείωσαν οι συντονιστέ σε δύο newsletters το 2 του Ιανουαρίου και 3 του Φεβρουαρίου αντίστοιχα 2013. Στα διάφορα αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου και τα σημεία που είναι εκεί στην ημερήσια διάταξη, δύο δηλαδή, θα συζητηθούν στις 18 και 19. Επαναλαμβάνω, 7 Μαρτίου δεν έχει Επιτροπή Μεταφορών ακυρώνεται η συνεδρίαση. Ματαιώνεται και τα σημεία που θα συζητούσαμε τότε θα συζητηθούν αργότερα στις 18 και 19 Μαρτίου. Για την εξυπηρέτηση εδάφους αποφάσισαν οι συντονιστές να στείλουν επιστολή στον πρόεδρο και να ζητήσουν τι γίνεται με τις τροπολογίες στην Ολομέλεια, ποιος δικαιούται να τις υποβάλει. Ε, γιατί ε, ε, οι συντονιστές συνιστούν να μην επιτρέπουν τροπολογίες στην Ολομέλεια. Λοιπόν, αυτά αποφάσισαν οι συντονιστές και σας τα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος. Είστε όλοι ευτυχείς με αυτά που ακούσατε. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα λίγο τσάι παρακαλώ. Και τώρα έλεγα Κανονικά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη που είναι η προσωρινή παρέκκληση από την οδηγία για ε, το ETS, το σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων εκπομπής αριού θερμοκηπίου εντός κοινότητας. Για στιγμή να πάρω λίγο το τσάι μου να ξυπνήσω, να πάρω δυνάμεις να προχωρήσω. Ah, oui, Can we check whether the system's working? Ελέγξουμε παρακαλώ αν λειτουργεί το σύστημα. Ε, αρχή της ψηφοφορίας, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Με χαρά. Ανακοινώνω ότι το ΕΛΚ δεν έχει υπερβολικά πολλούς που ψηφίζουν. Αυτό είναι κάτι νέο. Όλα καλά. Το ΕΛΚ έχει τις ψήφους που πρέπει. εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν συμβαίνει συχνά. Ε, αργότερα θα ακούσω μια ε, προφορική τροπολογία. Ο Ντίτερ, συγγνώμη δεν βρίσκω την κάρτα μου. Θα ακούσουμε ε, τις ψήφους, ε, θα σημειώσουμε τις ψήφους του κυρίου Κόχ, αρκεί να μην ξεπεραστεί το όριο ε, του ΕΛΚ. τροπολογία 6, Βίλς, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 23 κόκ και γκάλερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 φώστερ και λοιπά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 22, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Ο κύριος Κόχ είναι, ψηφίζει υπέρ, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, τροπολογία 24 και 16. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριε Ντεβεϊράκ, έχετε μια προφορική τροπολογία νομίζω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Right. That... not... Αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Δεν θέλετε να την ακούσετε πρώτα. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Δεν είναι δικαιολογία αυτό, Μάικλ. Κριστίν, μπορείς να την ε, διαβάσεις, αλλά υπάρχει αντίρρηση. Θες να προχωρήσεις? Θες να τη διαβάσεις. Ωραία, παρακαλώ να τη διαβάσεις και θα σημειώσουμε την ε, αντίρρηση που υπάρχει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως σα είπα χτε το απόγευμα θα ήθελα να υποβάλω προφορική τροπολογία για το θέμα που συζητήσαμε χτε το απόγευμα γιατί θεωρώ απαράδεκτο να υποστούν κυρώσει οι νομοταγεί. Αλλάζουμε τους κανόνες αλλά γιατί να πληρώσουν την ύφη νομοταγής. Έχω κάνει δύο τροπολογίες γραπτές 15 και 25 ε, για εταιρείε που έχουν λάβει διεθνεί πιστώσει, αφελώ, πιστεύοντα τα λεγόμενά μα και του επιτρόπους ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια φέτο. Άκουσα του συναδέλφου που λέγουν ότι θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε τρίτε χώρε και προτείνω λοιπόν ε, και θεώρησα ότι αυτό είναι συνενετικό. Μέχρι το τέλη του 2013 να επιτρέπεται και αν δεν βρεθεί συμβιβασμό για τις εξοκοινωτικές πτήσει, να επιτρέπεται στις εταιρείε μας να ε, χρησιμοποιήσουν αυτές τις πιστώσει ε, πριν καταστούν απόλυτε ζημίες. Ε, εάν δεν συμφωνείτε να τις αποσύρω. Σα είπα ε, ότι έχω αυτή την προφορική τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, η ε, ένσταση παραμένει, ναι, άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Πάμε λοιπόν στην αρχική τροπολογία 25 και την 15. Θα τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε παρακαλώ να ελέγξουμε τις δύο αυτές τροπολογίες, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας, ο κύριος Κοχ είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 ε, της κυρίας Πέρκερ. υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη only. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος είναι και η λέξη only, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 12 καταπίπτει. Ε, καταπίπτουν επειδή δεν υιοθετήθηκαν 21 και 23, η τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ τη 13, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Ο κύριος Κόχ είναι υπέρ, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. As everybody voted, Mr. Ψήφισαν όλοι, ο κύριος Κόχ υπερψηφίζει, λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, μία ψήφος κατά, 6 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Ε, συγχαρητήρια κύριε Γκρός. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η λεπτομέρειε τη επίτευξη του στόχου μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα. Έχουμε σχέδιο γνωμοδότηση. Ο κύριος Ρούμπιαλ. Ah, Συγγνώμη, κυρία Γκαριασά Ρουμπιάλ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Εδώ είμαι. Εγώ είμαι. Γκαρδιασάμπαλ με λένε βασικά. Ρουμπιάλ είναι το δεύτερο επώνυμο που έχουμε εμεί οι Ισπανοί, όπω γνωρίζετε. Έχουμε και το πατρικό και το μητρικό. Όλου του προγόνου του κουβαλάμε με επώνυμα. Εν πάση περιπτώσει, Γκαρδιασάμπαλ είναι το πρώτο. Ε, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Λέω κι εγώ ποιο είναι αυτό ο Ρομπιάλ. Ναι, ξέρω ότι είναι πιο εύκολο να το προφέρει από τον Καρδιά αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, Όπω έλεγε, γνωμοδότηση εμεί ε, παρουσιάζουμε στην πρόταση κανονισμού και θα ορίσουμε ε, τις προδιαγραφές για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για να φτάσουμε στο στόχο που γνωρίζετε ότι έχει τεθεί στα 95 γραμμάρια. Βεβαίως, το πρώτο είναι ότι επαναλαμβάνουμε αυτό το στόχο και το τονίζουμε, όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήταν έτσι και μια πρώτερη συμφωνία. Και τώρα, υπό το φως όλων των νέων στοιχείων και των αριθμών που έχουμε, Παραμένει αυτός ο στόχος φιλόδοξος πλην εφικτός. 95 ε, γραμμάρια μέχρι το 2020, διοξίδιο του άνθρακα εκπομπές. Έχω κάνει 20 τροπολογίες στον κανονισμό αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε τέσσερις βασικές ομάδες. Το πρώτο είναι ο στόχος μετά το 2020. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το εάν και κατά πόσο στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να βάλουμε στόχο για την περίοδο μετά το 20. Ξέρετε, επιχειρήματα υπάρχουν και υπέρ και κατά και πιστεύω ότι ευσταθούν όλα, έχουν ένα τμήμα ε, λογικής και δίκαιου, γιατί από τώρα δεν ξέρουμε μετά το 2020 τι τεχνολογία θα έχουμε, πώς θα έχει εξελιχθεί και πώς ε, θα είναι οι προδιαγραφές ελέγχου και μέτρησης ε, του διοξιδίου του άνθρακα και των εκπομπών του. Πάντως θεώρησα σημαντικό, αν μη τι άλλο, να μην βάλω συγκεκριμένο στόχο, αλλά μια κατεύθυνση να δώσω για το πού θέλουμε να πάμε και η αυτοκινητοβιομηχανία μετά το 2020. Διότι ποιο είναι το πρόβλημα αν δεν βάλουμε κανένα στόχο. Όπω γνωρίζουμε, ένα αυτοκίνητο δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται σχεδιασμό, ε, ανάπτυξη, τεχνολογία. Για να κυκλοφορήσει ένα μοντέλο χρειάζεται ένα ε, χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που κάποιος θα το συλλάβει μέχρι να κυκλοφορήσει στην αγορά μπορεί να περάσει και 8 ετία. Λοιπόν, αν δεν ξέρουμε μετά από το 2020 πού θέλουμε να πάμε από πλευράς εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αν δεν καταφέρουμε και συμφωνήσουμε, μετά το 20 όταν εκπνεύσουν οι στόχοι δεν θα έχουμε κανένα καινούριο. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ενδιαφέρον, αντί να βάλουμε συγκεκριμένο στόχο αριθμό, να βάλουμε ένα φάσμα δυνατοτήτων και για το 2025 ας πούμε να είναι 65 με 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές θα το έχετε διαβάσει, έχουν έρθει πολλά έγγραφα στόχος λοιπόν για το 2020 θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτή την ψαλίδα, βάση περιπτώσει 65 με 75 γραμμάρι. Το δεύτερο μεγάλο μπλοκ τροπολογιών που έχω καταθέσει έχει να κάνει με τις υπερπιστώσεις. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να βάλουν έτσι ένα πρίμα, ας πούμε, ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι ώστε οι κατασκευαστές που φτιάχνουν αυτοκίνητα που εκπέμπουν κάτω από 35 γραμμάρια ε, στην περίοδο από το 20 έως το 23 να επιβραβεύονται. Αυτά τα ονομάζουμε επιστοτικά υπερμόρια. Ε, να επιβραβεύονται λοιπόν οι εταιρείε που συνεχίσουν να επενδύουν στη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, αλλά με τη δική μας πρόταση όχι μόνο βελτιώνουμε και δίνουμε κίνητρα στη βιομηχανία, αλλά υπάρχουν και κυρώσεις. Και κυρώσεις δεν είναι για να τιμωρήσουμε τη βιομηχανία γιατί έτσι, αλλά ε, για να είναι στην Ευρώπη ε, η βιομηχανία μας ευθυγραμμισμένη με αυτά που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, που έχουν σύστημα και κινήτρων και κυρώσεων. Γιατί εμείς θα θέλουμε να μην ακολουθήσουμε ίδιο σύστημα περίπου με τις Ηνωμένε Πολιτείες, υπάρχει ένας κίνδυνος. Εκεί θα έχουν ε, ένα ελάχιστο στόλο που θα εκπέμπει κάτω από 35 ή 25. Ε, κινδυνεύουμε εμείς η παραγωγή να χαθεί από εμά. Αυτό που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας στην Ευρώπη. Τρίτη μεγάλη ενότητα τροπολογιών έχει να κάνει με τις παράμετρες χρηστικότητα, ε, παραμέτρους συγγνώμη, χρηστικότητας. Ε, θα είναι η μάζα ή το αποτύπωμα. Πώς θα το μετράς. Είναι δύο διαφορετικές τεχνικές. Αλλά πιστεύουμε ότι επειδή στο μέλλον το λογικό είναι ε, να χρησιμοποιηθεί μάλλον το αποτύπωμα, αρχίζουμε από τώρα να ανοίγουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή σε αυτές τις τροπολογίες τι κάνουμε, επιτρέπουμε απλούστατα ε, οι κατασκευαστές και οι ε, αντιπροσωπείες να αποφασίσουν αν θέλουν να χρησιμοποιούν ως παράμετρο χρηστικότητας τη μάζα ή το αποτύπωμα και να υπάρχει μέχρι το 2025 μία περίοδος προσαρμογής για να μπορέσουν όλοι να περάσουν στο αποτύπωμα. Και η τέταρτη μεγάλη ενότητα έχει να κάνει με τις αποκλήσεις όλες που έχουμε μεταξύ των εκπομπών που καταγράφονται τύπου ας πούμε και των πραγματικών εκπομπών. Γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ποιο είναι. Ένα τμήμα αυτών των μειώσεων δεν οφείλονται στη βελτίωση των αυτοκινήτων αλλά δεν συνάδουν τα πραγματικά στοιχεία με τα τυπικά που βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά όταν πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Και τελικά η κατανάλωση δίζελ ή βενζίνης ε, όχι μόνο είναι διαφορετική από αυτή που γράφει το αυτοκίνητο αλλά και οι πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν είναι οι αναγραφόμενες και εκείνες που υπόσχονται. Είναι υψηλότερε. Άρα δεν καταφέρνουμε να φτάσουμε στον πραγματικό στόχο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα εξού και κάποιες αρκετές τροπολογίες που κατευθύνονται προς τη βελτίωση και των μετρήσεων και ε, θέλουμε να βοηθήσουμε να αλλάξει ε, η διαδικασία δοκιμών, ο κύκλος δοκιμών, test cycle όπως το λένε. Και αυτό τον καιρό γίνεται συζήτηση και θέλουμε να έχουμε ένα έλεγχο πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο κοντινό στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάσταση των απολογιών λήγει την επόμενη Τρίτη για την γνωμοδότησή μου και μετά όταν θα λάβω όλες τις τροπολογίες θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμβαστικές έτσι ώστε η Επιτροπή μας να έχει θέση κατά πλειοψηφία για τη γνωμοδότηση αυτή. Αυτά και τελείωσα. Thank you very much. I've only got two shadows present at the moment, so I'll start with... Δύο σκιώδεις όλους και όλους έχουμε παρόντες. Θα μιλήσετε ε, εξ ονόμου του κύριου Φρός. Ναι, ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πολύ. Λόρες. Ήθελα να κάνω ε, κάποιες ε, προσωπικές παρατηρήσεις ε, μέχρι να καταφέρω ο Σκιώδης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά του και στην Επιτροπή μας, αλλά και στην γενική προοπτική το διοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει πάντα όμως να προσέχουμε στο θέμα αυτό. Να διασφαλιστεί η παραγωγή στην Ευρώπη. Και αυτή θα διασφαλιστεί με δύο τρόπους. Καταρχήν αν στηρίξουμε την ε, έρευνα και την ε, τεχνολογία ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να μην ε, θεσπίσουμε κριτήρια που να καταστήσουν αδύνατη την παραγωγή εντός της Ευρώπης. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε βρει καλή ισορροπία ανάμεσα αφενός στους στόχους και αφετέρου στις δυνατότητες της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με βρίσκει κάπως επιφυλακτικό διότι Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να εξετάσουμε και τι είναι δυνατόν σε ε, τεχνολογικό επίπεδο να κατά τη θέσπιση των στόχων μας δηλαδή να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω ε, έχει να κάνει με αυτά τα super credits. Ε, στην πρόταση της η, πρόταση της εισηγήτριας είναι κατά τη γνώμη πολύ καλύτερη από την πρόταση της ε, Κομισιόν. Πιστεύω ότι η αρχική πρόταση είναι υπερβολικά ισχνό κίνητρο. ώστε να ε, έχουμε άλλες ε, δυνατότητες ώστε να αναζητηθούν άλλες δυνατότητες. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει τα super credits ε, να ε, αποτελέσουν ανταμοιβή για τους παραγωγούς αυτοκινήτων. Αυτές ήταν οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Ελπίζω ο συνάδελφο Φλόρενς, που είναι σκιώδη εισηγητής, να μπορεί να πει περισσότερα. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχήν την εισηγήτρια τη δουλειά που έχει κάνει. Έχει ε, εργαστεί με μεγάλη επιμέλεια, το ακούσαμε αυτό, ε, όσον αφορά ε, τα μέτρα τα φιλικά προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να ε, τα προσέξουμε αυτό. Αναφέρθηκε και από την εισηγήτρια και από τον ε, κύριο Γκρόσο ότι θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική η βιομηχανία αυτοκινήτων της Ευρώπης. Ε, γι' αυτό όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν ήδη έχει προχωρήσει αρκετά με την πρότασή της και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις που να ξεπερνούν αυτήν. Καταλαβαίνω αυτό που λέει η συγγήτρια κυρία Ρουμπή, αλλά ότι θέλω να προχωρήσω και να υποβάλω και άλλες προτάσεις και να ε, υποδείξω την κατεύθυνση, αλλά κατά τη γνώμη μου ε, έχει πράγματι υποδεχθεί η κατεύθυνση και ε, ποιο ξέρει τι θα γίνει όταν αρχίσουμε να εξετάζουμε νέε παραμέτρου. Γι' αυτό διαφωνώ και νομίζω ότι μετά το 2020 ίσω να μην μπορούμε να θέσουμε καν στόχου. σε άλλου τομεί με την έρευνα και την τεχνολογία έχουμε δει εξελίξει που δεν τι περιμέναμε καθόλου όσον αφορά τα πιστοτικά υπερμόρια, τα super credits. Πάντα βρίσκω ότι είναι καλό να υπάρχει ένα ε, σύστημα κινήτρων, απλά θα πρέπει να φροντίσουμε το σύστημά μας ε, να ε, ανταποκρίνεται σε όλους τους βιομηχανούς αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Δεν έχουμε μόνο μικρά αυτοκίνητα, έχουμε και μεγάλα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην ε, ε, βρεθούν σε μειονεκτική θέση ε, όλοι όσοι παράγουν μόνο μεγάλα αυτοκίνητα. Πάντα είναι καλύτερα τα κίνητρα από τις ποινές, από τις κυρώσεις, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το σκεφτούμε. Όσον αφορά την παράμετρο χρηστικότητας, χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πάντα θα πρέπει να εξετάζουμε αν ε, αυτά που λέμε ε, αρκούν για να υπάρξει ε, διαφάνεια και σαφήνεια στον τομέα του διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνώ όσον αφορά τις Συμφωνώ γενικά. Όσον αφορά τι τροπολογίε, θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε, αλλά γενικά βρίσκω πολύ καλή την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο υποθέτω στο όνομα της κυρίας Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ε, λίγα λόγια ε, εκ μέρους της κυρίας Ρόσμπαχ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά που έχει κάνει πάνω στην έκθεση αυτή. Η σκιώδης εισηγήτρια συμφωνεί με την διόρθωση της διαφοράς ανάμεσα στις πραγματικές εκπομπές και σε αυτές που έχουν υπολογιστεί το ECR μπορεί να είναι διχασμένο όσον αφορά ε, την πρόταση του να έχουμε δύο ε, λύσεις όσον αφορά τους ε, στόχους για τα για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και και όσον αφορά τα όρια του διοξιδίου του άνθρακα, τα 35 γραμμάρια και δεν συμφωνούμε να θεσπίσουμε από τώρα στόχο για το 2025. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο τέλος του 2014 ε, να επανεξεταστεί η κατάσταση. Αυτή είναι η πρόταση της Αναρόσπαχ. Ευχαριστώ κύριε Στέιλερ ε, για τους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, για τη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Πρόσφατα συμμετείχα σε συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και ακούσαμε ότι οποιαδήποτε αποδυνάμωση στην πρόταση όσον αφορά τα γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα θα υποσκάψει τους στόχους μας, τους στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Όταν συζητάμε λοιπόν τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στο μέλλον, θα ήθελα να προτείνω αν ε, αντί να αποδυναμώσουμε τα μέτρα μείωσης, ενισχύσουμε τα μέτρα, τότε θα ε, αυξήσουμε τη μείωση διοξιδίου του άνθρακα, που νομίζω ότι είναι αυτό που προσπαθούμε όλοι να μας να πετύχουμε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι στόχοι που ε, προτείνονται 80 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο για τα αυτοκίνητα και 118 ε, για τα φορτηγάκια. Είναι και τα δύο επιτεύξιμοι στόχοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί. Είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη η λέξη αυτή στην πολιτική, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί και φιλόδοξοι όσον αφορά τον καθορισμό στόχων μέχρι το 2025, ώστε ο βιομηχανικός τομέας να ε, ε, ε, ξέρει που κινείται. Άκουσα επίσης ότι θα, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά και είμαι πεπισμένος ότι οι ίδιοι οι βιομήχανοι θα πρέπει να το κάνουν αυτό με βάση την αρχή ο πληρώνει. Βέβαια, οι βιομήχανοι οχημάτων ε, παρέχουν ε, ε, θέσεις εργασίας και καλύπτουν την ανάγκη για οχήματα. Απ' την άλλη, σε μια εποχή που κερδίζουν πολλά, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν θα πρέπει να φέρουν το κόστος της επίτευξης των στόχων. Εάν δεν πετύχουμε τις μειώσεις αυτές, τότε ο πλανήτης και όλοι όσοι βρίσκονται πάνω του που θα νιώσουν τις χειρότερες ε, ε, επιπτώσεις ε, της αλλαγής του κλίματος. Προσλέπω λοιπόν στη συνεργασία με την εισηγήτρια όσον αφορά τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε και προσλέπω και στην τελική ψηφοφορία. Κύριε Ζερίκε. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του. χαίρομαι η εισηγήτρια μας Χαίρομαι πολύ για το πρόγραμμα αυτό, γιατί νομίζω πως αυτή η σταδιακή προσαρμογή μέχρι το 2016 θα είναι πολύ ευφυής, γιατί ε, συνδυάζει το παρόν με το μέλλον και είναι προ, προνητική όσον αφορά τις δοκιμές των κατασκευαστών, γιατί όπως είδαμε και πριν από λίγες μέρες, αυτές οι δοκιμές εντείνονται για να προληφθούν τα προβλήματα. Ε, τώρα, για τον στόχο 2025. Ε, θα ήταν ε, επιθυμητό να πούμε ότι ναι, θέλουμε να προβλέψουμε τα όσα θα γίνουν το 2025, αλλά είναι περίπλοκο να δώσουμε αριθμητικά στοιχεία, γιατί βλέπουμε ότι ε, το άνοιγμα είναι μεγάλο, ενώ συζητάμε για 0,01. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να συζητήσουμε κατά πόσο θα δώσουμε συγκεκριμένα νούμερα ή όχι. Και μια τελευταία παρατήρηση για την οποία θα υποβάλω και τροπολογίες είναι ε, η κατανομή της προσπάθειας για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και για την κλίση αυτή η οποία αντιστοιχεί στα στοιχεία του 2006 ενώ τα στοιχεία τα επικυρωμένα για το 2009 υπάρχουν και θα πρότεινα να γίνει διόρθωση με τα πιο πρόσφατα στοιχεία γιατί αλλάζει για τα γεωταχή όχι αλλά για τα ελαφρά οχήματα ναι. Ε, αλλάζουν τα στοιχεία. Να ληφθούν υπόψη λοιπόν στους υπολογισμούς γιατί δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε πεπερασμένα στοιχεία. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν την ημερομηνία λήξης. Σας ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ησυχιατρία. Εννοείται πως όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε και να εξασφαλίσουμε την μείωση της ρήπανσης αλλά και του θορύβου που προέρχεται από τα οχήματα. Έχει γίνει καλή δουλειά μέχρι στιγμή. Αυτό το οποίο εμείς καλωσορίζουμε και αυτό προκύπτει, προέκυψε μάλλον από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν το ότι αποκλείονται πολύ μικρή παραγωγή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μικροί κατασκευαστές γιατί νομίζω αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Τώρα όσον αφορά την εισηγήτριά μας εδώ και τα όσα εμείς ε, μας απασχολούν στην Επιτροπή Μεταφορών θα, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν άλλοι σε σχέση με αυτόν τον στόχο του 2025 που δεν νομίζω πως είναι απαραίτητος, γιατί αυτό αφορά τους υπάρχοντες στόχους, δεν δημιουργεί καινούριου από όσο καταλαβαίνω. Και επίσης κάποιες τροπολογίες που έχουν τεθεί σε σχέση με την αξία αποτυπώματος. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε ισχύει κάτι τέτοιο, ε, αν δώσουμε μια αξία αυτή τη στιγμή. Κάποιες τροπολογίες μπορούμε να τις στηρίξουμε εύκολα, αλλά κάποιοι από εμά έχουμε... Βλέπουμε μεγάλες διακοιμάσει στην αυτοκινητοβιομηχανία στις περιφέρειές μας και σίγουρα θα στηρίξουμε κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για να θέσει σε κίνδυνο την αυτοκινητοβιομηχανία. Περνάνε πολύ δύσκολους καιρούς και πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους και σαφείς στόχους και αυτό θα σκοπεύω να κάνω. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Μπέργκερ. Λίχτεμπέργκερ. Ευχαριστώ. Όταν ακούω πάντα ρεαλιστική στόχη και ευελιξία, αρχίζω και ενδιαφέρομαι για τον εξή ειδικό λόγο. Σε τελική ανάλυση, αυτά είναι συγκάλυψη για να μην κάνουμε αυτά που αποφασίσαμε βάσει επιστημονικών αναλύσεων και προσπαθούμε κάθε νομοθεσία ή κάθε υλοποίηση των όσων έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ε, ε, με μεγάλη βιβλιοψηφία να την καταργήσουμε. Και θέλω να τονίσω, και δεν είναι προς όφελος όλης της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά ενός και μόνο τμήματος και ένα τμήμα που δεν θέλει να αλλάξει τακτική και δεν θέλει να προσαρμοστεί. Γενικά δεν είναι ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία αυτή γιατί υπάρχει και ο καινοτόμο τομέα στη βιομηχανία και κάποιου άλλου που θέλουν να κάνουν 15 βήματα πίσω, όχι ένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε όλους αυτούς να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι και αν θέλουμε να συνεχίσουμε ε, με ε, ε, την παλιά τακτική. Ξέρετε το παλιό παιχνίδι το Μικάντο, όποιος κινείται πρώτος έχασε δεν θα πετύχουμε κανένα στόχο. Ε, αν θέλουμε να μείνουμε σε αυτές τις αγκυλώσεις και την ακινησία. Και σήμερα τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, επιτέλους, αργά, αργά, αργά, αλλά σταθερά δημιουργείται ε, και η επίγνωση ότι ξέρετε αλλάζει το κλίμα και μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το καταπολεμήσουμε. Και βέβαια είναι και κάποιοι άλλοι που θέλουν να αγοράσουν κάτι καρακουρσάρες για να κάθονται μπλοκαρισμένοι στα ποτηλιαρίσματα. Αλλά αυτό θέλουμε. Εμείς σε αυτούς θα προσανατολίσουμε την πολιτική μας για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Αυτοί θα κανονίζουν τι θα γίνεται. Πρώτον, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί το καινοτόμο τμήμα τη αυτοκινητοβιομηχανία καθίσταται μονίμω όμοιρο για εκείνου που δεν θέλουν να το κουνήσουν ρούπι και θέλουν να επιστρέψουν ε, νομοθετικά και πίσω από την κατάσταση του 1990 στην πρώτερη κατάσταση. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να επιβραβεύσουμε τους καινοτόμου και τους νεοτεριστές και τους πρώτοπόρου. Ναι λοιπόν στο στόχο του 2020 ε, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με την αξιοπιστία μας να κάνουμε πάντα ένα βήμα μπρος και δύο πίσω και Μην βάζουμε τέτοια συνθήματα και τέτοιες λέξεις που επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Αν αρχίσουμε την ευελιξία και στο ποινικό δίκαιο, ε, αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα για την επιβολή της νομοθεσίας. Και κάτι με το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ είναι οι πραγματικές τιμές και αυτή η ιστορία. Βλέπουμε τώρα ε, στα φορτηγά ότι απέχουν έτη φωτός οι πραγματικές μετρήσεις από εκείνες ε, που γράφουν τα συνοδευτικά έγγραφα και η περιγραφή του οχήματος θα πρέπει όλα αυτά να προσαρμοστούν, να ευθυγραμμιστούν. Ε, τεχνικά δεν είναι και καμιά τεράστια πρόκληση. Αυτά είναι μπανάλ πράγματα καθημερινά. Κύριε Σαουβάρμα. uh, Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σκληρή της δουλειά και οι παρατηρήσει τη κυρία Λίχτενμπεργκερ με οδηγούν στο να πω τα εξή. Κάθε φορά που ακούω εγώ τι λέξει επιστημονικά στοιχεία κυρίως συνδυαζόμενα με τη φράση και παραθέτω εάν δεν ενεργήσουμε τώρα τα παιδιά μας το χρόνο, το έτος τάδε δεν θα έχουν πια το πλανήτη ε, έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα με το να αναγκάσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία να, να αποδώσει καλύτερα βελτιώνοντας τις ε, αποδόσεις των αυτοκινήτων ε, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Αλλά ας είμαστε λογικοί. Ε, ε θέλω να είμαστε λογικοί. Δεν είμαι ε, φανατικός, αλλά ας είμαστε λογικοί. Ας δούμε άλλα δύο χρόνια. Συμφωνήσουμε με τον για ένα-δύο χρόνια και μετά να ξαναδούμε τι, τα στοιχεία που θα έχουμε. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες με αυτή την προοπτική. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματο της Κομισιόν, ο κ. Χότζον από την Γενική Διεύθυνση ε, ε, κλιματικών αλλαγών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να αναφερθώ στα τέσσερα σημεία που θέτει η εισηγήτρια. Για το θέμα των δοκιμών, το κύκλο δοκιμών, η Κομισιόν συμφωνεί ότι σίγουρα ο καταναλωτής χρειάζεται πιο ακριβείς πληροφορίες και, συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους για ε, μια διαδικασία τέτοιου ελέγχου. Πιστεύουμε πως οι τροπολογίες που έχουν γίνει και οι βελτιώσεις στη διαδικασία θα οδηγήσουν σε πιο ακριβή αναφορά ε, για τις εκπομπές. Λοιπόν, ε, ε, για το θέμα των εκπομπών το βρίσκουμε δύσκολο να θέσουμε όρους. Ε, αναγνωρίζουμε την αλλακτική λύση ότι είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ότι δίνει στους κατασκευαστές το κίνητρο να επιτύχουν φιλόδοξες πωλήσει Τόσο έχουμε εκτιμήσει και τον αντίκτυπο των διαφόρων καθεστώτων που προτείνονται και ο αντίκτυπο ε, διοξιδίου του άνθρακα αυτή τη προσέγγιση θα είναι μικρότερο ε, αντί για το καθεστώ των σούπερ πιστώσεων ε, όπου συμμετέχουν διάφοροι πολλαπλασιαστέ. Τώρα, όσον αφορά το αποτύπωμα, έχουμε σκεφτεί αρκετά αυτό το θέμα του αποτυπώματο στην προετοιμασία αυτή τη πρόταση. Θα ήταν σωστό να πούμε πω αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφέ ποιε θα ήταν οι καλύτερε παράμετροι και έχουμε ενδείξεις πως το αποτύπωμα φαίνεται να είναι φθηνότερος τρόπος κάπως για να πετύχουμε μειώσεις του διοξιδίου, αλλά και πάλι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους κατασκευαστές. Βλέπουμε ωστόσο κάποιες προκλήσεις εάν εισαχθεί διπλό σύστημα και ήδη έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Για το θέμα τώρα μετά το 2025 και τους πιθανούς μελλοντικούς στόχους. Ε, το εύρος που προτείνεται είναι αρκετά φιλόδοξο όσον αφορά το ποσοστό μείωσης και είναι ψηλότερο από αυτό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η μελέτη μας δείχνει πως είναι εφικτό πάνω κάτω με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, αν και θα σήμαινε αυτό ε, σημαντικά επίπεδα υβριδισμού αυτό ούτω ή άλλω το επιδιώκουν οι περισσότεροι κατασκευαστές και είναι πιθανόν από την εκτίμηση της ε, Κομισιόν να δούμε ότι ο στόχος των 70 γραμμαρίων είναι ε, εφικτός. Ε, θέλει η συγγήτρια να απαντήσει. Θέλω, ευχαριστώ πολύ, Μπράιν, πάρα πολύ σύντομα, γιατί όπως είναι διαφορετικές οι θέσεις ανάλογα με την πολιτική ομάδα στην Επιτροπή μας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με τους στόχους ε, το 2020 ε, και μετά το 2020 μάλλον. Αυτό είναι από τα πιο επίμαχα σημεία. Και πολλοί ε, μίλησαν για λογική, για ισορροπία, για αναζήτηση λίγο ισορροπίας μεταξύ εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αυτού που θέλουμε όλοι που είναι η μείωση, αλλά να σκεφτούμε και τη βιομηχανία και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε στην Ευρώπη την παραγωγή αυτοκινήτων. Μα γι' αυτό το λόγο προτείνω ε, αυτή την ψαλίδα, αυτό το φάσμα 65 με 75 δεν είναι ένα το γραμμάριο, ε, σας δίνει ένα περιθώριο 10 γραμμαρίων γιατί δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία για το τι θα γίνει μετά το 2020 και πού να ξέρουμε. Γι' αυτό βάζουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ψαλίδα ας πούμε, και το μεγάλο περιθώριο για να δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος που θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μετά το 2020 με κίνητρα για να ξέρει και η βιομηχανία που κινείται και συμφωνία άλλωστε και ίδια. Αυτοί οι πρώτοι είναι εκείνοι που επενδύουν. Έτσι δεν είναι, για να μειωθούν ε, οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Πάντως είναι γεγονό ότι τα στοιχεία δεν τα έχουμε ακόμα για το, μετά το 2020. Και λογικό θα ήταν να πει κάποιο ότι δεν έχουμε την ε, πληροφόρηση, α περιμένουμε. Το πρόβλημα είναι πόσο θα περιμένουμε, γιατί όπω σα είπα, αν μέχρι το 2018 δεν έχουμε ε, μόνιμη, βάσιμη ε, πληροφόρηση και ε, αξιόπιστη, δεν μπορεί η βιομηχανία να φτιάξει αυτοκίνητα για μετά το 2020. Για να βγει ένα αυτοκίνητο στην αγορά από τη σύλληψή του χρειάζεται 7-8 χρόνια να γεωτοχεί και 10 χρόνια τα εμπορικά οχήματα, τα επαγγελματικά. Ε, λοιπόν, Γι' αυτό βάζουμε αυτό το στόχο που είναι και φιλόδοξος αλλά και ευρύς για μετά το 2025. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αυτοκινητοβιομηχανία ε, από σήμερα μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια συμφωνήσουν για τους νέους στόχους και τη νέα μορφή και τρόπο μέτρησης στο διοξιδίου του άνθρακα, εξαφανίζεται αυτός ο κανονισμός και αντικαθίσταται από ένα καινούριο που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κληθεί και πάλι το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα μια ασφάλεια. Αν σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν χρειάζεται μια πρόταση του Κοινοβουλίου να υπάρχει, μπας περίπτωση. Αλλά είναι βρία, δεν είναι πολύ στενή. Και έχουμε δώσει μια κατεύθυνση. Αν έρθει νέα πρόταση, αν έρθει η αυτοκινητοβιομηχανία, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και συμφωνήσουμε για τους στόχους που θα είναι σαφείς για μετά το 2025, εξαφανίζεται αυτό παίρνουμε τα μέτρα μας, αν θέλετε, προ, τις προφυλάξεις μας. Κάτι προτείνουμε, αν δεν υπάρξει καμία συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένω τις τροπολογίες σας και ε, θα προσπαθήσω να κάνω συμβιβασμούς για να συγκεράσω τις διάφορες απόψεις και να έχουμε όσο γίνεται ευρεία πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να... Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι η τροπολογία για τις προθεσμία της τροπολογίας είναι 26 Φεβρουαρίου, μια εβδομάδα από σήμερα και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει μάλλον τον Απρίλιο 24-25 για τα αυτοκίνητα και 6-7 ε, Μαΐου για τα ελευθερά επαγγελματικά οχήματα. Πάντως δική μας ε, προθεσμία είναι 26 Φεβρουαρίου ε, και 26 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Να προχωρήσουμε στο επόμενο ε, θέμα στη Μέση διάταξη που θα, πραγματοποιηθεί και, θα συζητηθεί και κλεισμένων των θύρων. Παρακαλώ λοιπόν ε, να αποχωρήσουν όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής μας ε, και να καλέσουμε τον κύριο Γκουντρού.